Ε, κηρύσουν καινή τη θέση αυτή από 16 Ιουλίου 2010. Φάση του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στη συνάντησή της, της 5ης Ιουλίου 2010 επαλήθευσε τα διαπιστευτήρια των κύριων Μπέλα Κόβαξ από 31ης Μαΐου 2010 και της κυρίας Ιλντίκο Γκαλπελές και του κυρίου Κιθ Τέιλορ από Δευτέρα Ιουνίου 2010 και του κ. Λούκα Χάρτο και του κ. Γιάν Μέλντερ από 22 Ιουνίου 2010. Οπότε προτείνω να επιβεβαιωθούν οι εντολέ αυτές, να εγκριθούν. Σχόλιο παρακαλώ. Άρα εγκρίνονται οι εντολέ των ευρωβουλευτών αυτών. Τα πρακτικά θα πάνε για έγκριση στο Σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή τη